Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας ημέρα. Κύριε Λούντγκριν, θέλετε κάτι να μου πείτε. πρέπει να πω κάτι και παρακαλώ να είστε ήσυχοι και να με ακούσετε. Ξέρετε κάτι, πολλοί από εμάς σηκωνόμαστε έγκαιρα και περιμένουμε εδώ πέρα ότι θα αρχίσει η ψηφοφορία, είμαστε πέντε λεπτά πριν και περιμένουμε. Και είμαστε ήδη ε, πέντε λεπτά, μάλλον έρχεται η πρόεδρος πέντε λεπτά αφού έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι ψηφοφορίες και τρώει το πρωινό της και εξακολουθούν κάποιοι να έρχονται. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό, δεν είναι δείγμα σεβασμού και είναι και αλαζονικό όταν εμείς έχουμε έρθει εδώ. Εννέα η ώρα δεν υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινήσει η συνέντευξη και η ψηφοφορία. Δεν μπορείτε να έρχεστε εσείς 9 και 10 δεν είναι πραγματικά δείγμα σεβασμού. Κύριε Λούντγκρεν, σημειώνω την παρατήρησή σας. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσως. Παρακαλώ μήνυμα από τους διερμηνείς. Βρισκόμαστε στην 17η μέρα των κινητοποιήσεων και δεν έχουμε δει ακόμη καμία αντίδραση εκ μέρου τη διοίκηση. Ω εκ τούτου, σα πληροφορούμε με τα λύπη ότι η συνδιερμηνία θα σταματήσει ακριβώ στην προβλεπόμενη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Έχετε μέχρι τις, ε, σήμερα το μεσημέρι, λέει πρόεδρο, για να δεχθείτε τι προτάσει των συντονιστών. Nous avons un message des... Πριν ξεκινήσουμε, λέει η πρόεδρο, έχουμε να μην του διερμηνήσει. Βρισκόμαστε στη 17η μέρα των κινητοποιήσεων και ακόμα δεν έχουμε δει καμία αντίδραση εκ μέρου τη διοίκηση. Ω εκ τούτου, σα πληροφορούμε με τα λύπη ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ την προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση, δηλαδή στι 12.30. Ευχαριστούμε πολύ του διερμηνείς μα. Το ακούσατε. Θα πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο. Διότι και ο χρόνος είναι χρόνος. Προς σεβασμό λοιπόν, απέναντί τους δεν θα έχουμε διερμηνία μετά τις 12.30. Ευχαριστούμε. Ξεκινούμε με τις ψηφοφορίες. Δικαιώματα και υποχρεώσει των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών. Αναβλήθηκε αυτή η ψηφοφορία σε μελλοντική ε, ημερομηνία. Και περνάμε στην έκθεση ΟΕΛΗ. Η Ευρώπη σε κίνηση, θεματολόγια τη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινούμε αμέσω. Πρώτα απ' όλα να δούμε ότι λειτουργούν οι κάρτε και αν έχουμε αρκετέ παρουσίε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Allez, le vote est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. πολύ καλά αρκετούς σοσιαλιστές, αρκετούς ε, ΕΛΚ, αρκετούς ε, οικολόγους, αρκετούς ΑΛΔΕ έχουμε. Ξεκινάμε. Συμβαστική πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Μάλλον, συγγνώμη, 20. Συμβαστική 2. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Τροπολογία μάλλον 26. Επερ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, συγγνώμη, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε για την 40 άρχια την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική έξω Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε για τη 43. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 50. πέρας. Εγκρίνεται. Μάλλον απορρίπτεται. Ήταν για να δω αν έχετε ξυπνήσει. Είστε αρκετά ξύπνοι Τροπολογία 50 λοιπόν απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές να ελέγξουμε. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Ένβη 12. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ένβι 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. 87 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Αποχές. Απορρίπτεται. Envy 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28. 26 με συγχωρείτε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 20 υπέρ. Κατά αποχές Ένβι NV22 υπέρ κατά αποχές εγκρινεται ΕΝΒΙ NV16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβι 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές να ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 132. Πέρας. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. 133 κύριε Βαντενκάμπ. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά.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 Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα τελική ψηφοφορία. Άρχεται η τελική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Πέρας της ψηφοφορίας Η έκθεση εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Voilà. But ah, we don't have Mr. rapporteur.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 ο εισηγητής μας έχει φτάσει. Ισμαήλ, είσαι εσύ ο εισηγητής τότε. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Επανερχόμεθα λοιπόν. Λοιπόν, φτάνουμε στην παρουσίαση της Επιτροπής γύρω από την πρόταση δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Comme vous le savez, dans son discours... Όπως γνωρίζετε, στην ομιλία του το 2017 για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος Juncker προτείνει την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης στον κοινωνικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ομοθετική της πρόταση την άνοιξη του 2018. Η αρχή αυτή μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των κοινωνικών των κανόνων και στον τομέα των μεταφορών στον τομέα της απόσπασης των οδηγών, του χρόνου εργασίας, του χρόνου οδήγησης, του καμποτάζ. Είναι θέματα σημαντικά τα οποία ανήκουν στο πακέτο κινητικότητας επί του οποίου πολύ πρόσφατα ψηφίσαμε. Για τον λόγο αυτό λοιπόν η Επιτροπή μας έχει ξεκινήσει να εμπλέκεται στην ε, ε, πρόταση αυτή και θα γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή Εργασίας η οποία είναι φυσικά αρμόδια επί της ουσίας. Σήμερα θα ακούσουμε μια παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε 10 λεπτά έτσι ώστε να μας παρουσιάσετε τους άξονες εργασίας, κύριε Λιεζουά, και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ το Ισμαήλ. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Αυτή είναι μια αρχική πρόταση η οποία ανήκει στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο για την ολοκλήρωση όχι απλά της ευρωπαϊκής αγοράς αλλά μιας δίκαιης εσωτερικής αγοράς που σέβεται την εργασία. Έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Έχετε στην διαφάνεια αυτή αρκετά παραδείγματα. Άλλο παράδειγμα είναι και η αναθεώρηση των ομάδων συντονισμού για την κοινωνική ασφάλιση. Καθορίζονται λοιπόν οι βασικές αρχές στα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για σωστά λειτουργούσες αγορές εργασίας. Το θέμα της κινητικότητας είναι ένα βασικό θέμα βέβαια για να μπορέσω να παρουσιάσω περιληπτικά με λίγα λόγια την πρότασή μου θα χρησιμοποιήσω τη λέξη επιβολή. Νομίζω ότι η λέξη επιβολή είναι η βάση του πακέτου που ε, προτείνει τελικά την δημιουργία της αρχής ε, για θέματα εργασίας που θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση της επιβολής των, των κανόνων που ισχύουν στη φάση αυτή. Δεν θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της διασύνοριακής κινητικότητας. Το 2017 υπήρχαν πάνω από 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους που εργάζονται σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα προέλευσης. Η κινητικότητα λοιπόν έχει αυξηθεί από το 2007 μέχρι το 2017 κατά 65%. Έχουμε λοιπόν μια νομοθετική πρόταση για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής, ε, μιας εξωτερικής υπηρεσίας λοιπόν. Αν δείτε την πρόταση κανονισμού χρηματοδότησης, βασίζεται στις ε, βασικές αρχές οι οποίες ε, ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 για τις εξωτερικές υπηρεσίες, τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Επιτροπής, της Ένωσης μάλλον. Και υπάρχουν διάφορα άρθρα 48, 53, 62 που αναφέρονται στα θέματα της ελεύθερης διακίνησης, την διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης και φυσικά και το 91 για θέματα μεταφορών. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει μια σαφής αγκύρωση των μεταφορών στις προτάσεις για τη δημιουργία της υπηρεσίας ελέγχου εργασίας. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να καθορίσουμε το πεδίο ενασχόλησης της καινούργιας αυτής υπηρεσίας που δεν περιορίζεται μόνο στις διασυνοριακές μορφές απασχόλησης αλλά περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες στο ιδρυτικό της καταστατικό και άλλες πρωτοβουλίες. Αν βλέπετε τις λεπτομέρειες της πρότασης θα δείτε σαφείς αναφορές και στη μεταφορά, ιδιαίτερα στο άρθρο 71 με βάση τη κοινωνική νομοθεσία και θα υπάρξει και μια λέξη specialis ειδική στο μέλλον για τα θέματα της κινητικότητας και απόσπασης εργαζομένων. Τώρα, βασική στόχη της αρχής αυτής, ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και σωστή εφαρμογή των κανόνων που είναι σε ισχύ, έτσι ώστε να υπάρχει μια σαφής κατανόηση από πλευρά των εργαζομένων, των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεων. Δεύτερον, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών στα πλαίσια του πακέτου Mobility 1, Ας περάσουμε λοιπόν τώρα γρήγορα στις, στις δράσεις, στην αποστολή, στις αποστολές εισαγωγικά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε, ένα πρώτο προκαταρκτικό σχόλιο, η αρχή δεν θα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών επιβολής. Αυτό παραμένει ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίσουν την επιβολή, αυτό ισχύει σήμερα, αυτό θα ισχύει και για το μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η βασική αυτή αρχή θα είναι εκεί για να συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών. Δεύτερον, παρατήρηση δύο που μπορεί να είναι και αντικείμενο κριτικής από πλευρά σας. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα είμαστε επιτυχείς αν επιβάλλουμε την συνεργασία ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία της προσπάθειας. Λοιπόν, τώρα για την πρόσβαση στη σωστή ενημέρωση. Τι σημαίνει αυτό για τις οδικές μεταφορές. Ένα παράδειγμα. Μπορούμε να συλλέξουμε λοιπόν στον τομέα των οδικών μεταφορών λεπτομέρειες ε, για τις διάφορες χώρες και επίσης να ε, συντάξουμε και κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή εφαρμογή των προβλέψεων αυτών. Όπως επίσης και μια μόνο απευθυντική θηρίδα για τις ε, οδικές μεταφορές. Ε, ELA would provide operational support to national authorities. Again, what can that mean for road transport? ELA could, for example, promote... Λοιπόν, εμείς θέλουμε να προτείνουμε την ε, ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις εθνικές αρχές επιβολής και στην ψηφιοποίηση η οποία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για την επιβολή και η Ευρωπαϊκή Αρχή θα μπορούσε να ε, βοηθήσει ιδιαίτερα. Ε, μια τρίτη αν θέλετε βασική δράση είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των δράσεων στον τομέα της επιθεώρησης, του ελέγχου. Έχουμε αυτή τη στιγμή οργανώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έξι συντονισμένους τύπους μορφές ε, ελέγχων. Και εδώ η υπηρεσία θα μπορούσε να παρέχει τις απαιτούμενες ε, διευκολύνσεις γι' αυτό ταυτόχρονα και ανάλυση ε, και αξιολόγηση των κινδύνων για θέματα διασυνοριακής κινητικότητας ε, του εργατικού δυναμικού, όπως επίσης και ε, ενίσχυση των εθνικών αρχών μέσω σωστής συνεργασίας και αμοιβαίας καθοδήγησης. Και έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ισχύουσες διατάξεις. Το λεγόμενο capacity building. Βλέπουμε ότι ε, μπορεί να υπάρχουν μειώσεις της, στο, εργατικό, στο εργασιακό δυναμικό το οποίο αναφέρεται και ασχολείται με θέματα ελέγχων στον τομέα της εργασίας. Επίσης ε, διαμεσολάβηση, διαιτησία όταν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και στα θέματα τώρα της διακυβέρνησης, δύο είναι τα βασικά θέματα. Ποιοι θα είναι οι πόροι της αρχής όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε 144 υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων εθνικών υπαλλήλων και ένα προϋπολογισμό 51 εκατομμυρίων ευρώ και συμμετοχή φυσικά των κοινωνικών εταίρων. Είμαστε αισιόδοξοι σχετικά με την δημιουργία της υπηρεσίας αυτής. Ήδη έχουμε προβλέψει έναν προϋπολογισμό για το 2019 και νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν με ικανοποιητικό ρυθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την συστηματική συμμετοχή των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων αυτό σημαίνει λοιπόν θα έχουμε μια ομάδα με έξι αντιπροσώπους από τα συνδικάτα, από τους κοινωνικούς εταίρους, από τις επιχειρήσεις επίσης. Θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και φτάνω στην τελευταία διαφάνεια της παγουσίασής μου. Όλοι γνωρίζουμε ε, ότι η πρόταση έγινε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 13η Μαρτίου. Επίσης ε, πέρασε από το ΕΠΣΚΟ Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στις 21 ε, ή μάλλον σήμερα ουσιαστικά. Ε, υπάρχει επίσης ξεκινήσει η μαλλον σημερα ουσιαστικα υπαρχει επισης ξεκινησει η δουλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον εισηγητή σας, τον κύριο Λέναρς, και σκοπεύετε να ψηφίσετε το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ώστε να περάσουμε στην ψηφοφορία στον Ολομέλεια πριν το τέλος του 18. Εμείς θα θέλαμε να υιοθετηθεί η πρόταση στα πλαίσια της παρούσης κοινοβουλευτικής εντολής. Έχουμε, όπως είπα, δεσμεύσει ένα ποσό για τον προϋπολογισμό του 19 για να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας του ELA, του ELA, φιλοδοξία της Αυστριακής Προεδρίας είναι να καταλήξουμε σε μια γενική θέση. Ήδη έχουμε καθορίσει μια ομάδα συμβουλευτική η οποία δεν είναι ο χώρος διαπραγμάτευσης της πρότασης αυτής, αυτό θα το κάνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο στόχος όμως αυτής της διαπραγματευτικής ομάδας είναι να προπαρασκευάσει όλες τις επιμέρους ε, δράσεις της ε, νέας αυτής προτινόμενης αρχής. Αυτά. That's it. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις αντιδράσεις σας και να δώσω και απαντήσεις στο μέτρο του δυνατού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λιεζουά. Ξεκινά λοιπόν η συζήτηση αυτή αμέσω τον κύριο Σμέλερ Τούγκ, που αντικαθιστά τον εισηγητή μα, ο οποίο δεν μπορεί να είναι εδώ. Έχετε το λόγο, κύριε Τούγκ. Καλημέρα σα, ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητή είναι ο συνάδελφο Μίχαλ Ντέτχεν, ο οποίο δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει από σήμερα εδώ, οπότε θα παρουσιάσω εγώ το έγγραφό του στα γερμανικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν. Α, ναι, στα γερμανικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να πω τα εξή, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα ο συνάδελφος ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα και να παρουσιάσει ε, το έγγραφό του στην Επιτροπή Μεταφορών, διότι πρέπει να μιλήσει σε μια διάσκεψη για το θέμα κοινωνική Ευρώπη. Όμως, επί της ουσίας, θέλουμε ε, να συζητήσουμε την κοινωνική Ευρώπη, αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή και πώς μπορούμε εμείς στην εσωτερική αγορά να έχουμε πιο δίκαιες συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση τον Σεπτέμβριο τη προηγούμενη χρονιάς ήδη ε, είπε γιατί υπάρχει μια εποπτική αρχή για τις τράπεζες ε, που επιτηρεί την κατάσταση των τραπεζών και δεν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ε, για την ε, επιτήρηση των συνθήκων εργασίας. Έκανα αυτή τη σύγκριση και νομίζω ότι εμείς, Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών και με την Επιτροπή Απασχόλησης είναι καλό να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να συζητήσουμε και τις διάφορες απόψεις που ήδη προέκυψαν από τη συζήτηση για το πακέτο για την κινητικότητα. Πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση για τα, εκατομμύρια, ε, για τα πολλά εκατομμύρια ε, ανθρώπων που μετακινούνται. Βλέπουμε όμως μέχρι στιγμής οι νόμοι να μην έχουν φέρει τις απαραίτητες βελτιώσεις ε, και νομίζω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προωθήσει. Ε, τη βελτίωση δηλαδή της εφαρμογή της νομοθεσίας και εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το δικό μας ε, λιθαράκι γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσει, όπως παραδείγματο χάρη για τις διάφορα εργοτάξια, οι έλεγχοι δηλαδή που πρέπει να γίνονται στη οδική ασφάλεια κτλ. Οι εθνικοί επιχε... θεωρητές έχουν δεμένα τα χέρια σήμερα ε, όταν η έδρα παραδοσιακά τη εταιρεία είναι σε μια διαφορετική χώρα, έχουμε τις εικονικέ αυτέ εταιρείε, τι εταιρείε γραμματοκιβωτίων που ε, ουσιαστικά διαφεύγουν των μηχανισμών ελέγχου ε, και εκμεταλλεύονται τις ε, ιδιαίτερε μισθολογικέ συνθήκε, εργασιακέ συνθήκε των κρατών μελών. Εμεί θέλουμε να υπάρξει βελτίωση των εθνικών αρχών, να υπάρχει επαφή με όλους τους ενδιαφερομένους και οι εργαζόμενοι στο οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους. Ε, ε, το πρόβλημα των εργασιακών συνθήκων των οδηγών είναι πολύ σχηδή και πιστεύω ότι αυτή η εργασιακή αρχή θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό με βασικό καθήκον να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων ε, των εθνικών αρχών που δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση αλλά να υπάρξει μια συνεργασία ώστε Τώρα, να λάβουμε υπόψη στην έμπλα ε, της απόψης της ΤΡΑΝ, έχουμε ένα πολύ καλό ε, χρονοδιάγραμμα. 6 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας θα κατατεθεί το σχέδιο, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 12 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, στις 9 ε, Οκτωβρίου. Ο εισηγητής θέλει να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της ΔΕΛΤΑ ΜΟΥΒ και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Μεταφορών, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λουκασένσκα. Έχει τώρα το λόγο. Να σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που μου αρέσει είναι η συντομογραφία. Ε, έλα λέγεται αυτό, είναι Ευρωπαϊκή Αρχή. Έτσι με λένε και εμένα, έλα. Και ελπίζω ότι όσοι χρειάζονται πληροφορίες θα μπορούν να τις λάβουν από αυτή την εταιρεία, ότι αυτή ή από τη από αυτή την αρχή, η οποία θα υποστηρίζει πάντοτε την ενιαία αγορά, την αρχή της κινητικότητας και θα διασφαλίζει, θα προσπίζει τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού λοιπόν και θεωρώ ότι πράγματι είναι ανάγκη η δημιουργία της Ευρωπαϊκής αυτής αρχής εργασίας και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και πολιτική απόφαση. Ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι της Κομισιόν, Πρόσφαση στην πληροφόρηση, δημιουργία ψηφιακής πύλης, κατάρτιση, διαβούλευση, υποστήριξη των εθνικών αρχών. Όλα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. Πολλοί επιχειρηματίες αλλά και ελεγκτές αναζητούν ε, πληροφορίες ε, και στοιχεία για την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπεται στα κρατη Τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρχουν καταχρήσεις της νομοθεσίας και αποφυγή των προστήμων. Συνεπώς λοιπόν έτσι θα καθοριστούν οι ρόλοι της υπηρεσίας. Δεν θέλω να επαναλάβω εδώ αυτά τα οποία υπόθεσαν. Ε, φοβάστε ότι μπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις. Ε, δεν είναι μια υπηρεσία η οποία μπορεί να θίξει τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές και θα μπορούσε να μας πει η Επιτροπή που προβλέπεται να γίνει η, η έδρα της υπηρεσίας. Έχετε επιλέξει τη χώρα ή θα μπορέσουν οι διάφορες χώρες να διεκδικήσουν την εγκατάστασή της. Λοιπόν, στην ουσία περιμένουμε λοιπόν την τελική σας πρόταση. Θέλουμε να δούμε τι συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση αυτή και θα υποβάλουμε τροπολογίες. Αν πράγματι δημιουργηθεί με σωστό τρόπο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την αγορά εργασίας και τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους. Ευχαριστούμε κυρία Λουκασένσκα, ο κύριος Ζλωτόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι κάπως πιο επιφυλακτικός από τους προηγούμενους ομιλητές. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει κάποιο είδους ε, αστυνομία της απασχόλησης. Εάν τα κρατη πρέπει να ε, φροντίσουν για την εφαρμογή του νόμου ούτως ή άλλως, δεν χρειαζόμαστε μια ακόμα νέα αρχή που έχει αρμοδιότητα και πάλι να φροντίζει για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την αρχή όταν συζητήσαμε ανάλογα θέματα και είχαμε αναφέρει την ε, πιθανότητα δημιουργίας της. Η αρχή αυτή δεν έχει ακόμα ε, συσταθεί δεν ε, θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει βάση για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού στα πλαίσια της ε, επικουρικότητας. Όλα τα ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές ε, διευθετώνται στα επίπεδα των κρατών μελών και υπάρχει και στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, το ανέφερε και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει ανάγκη η νέα αρχή να οργανώσει τη συνεργασία, διότι υπάρχει ήδη. Έχουμε παρακολούθηση τη εργασία και τη απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλουμε λοιπόν να αποποιηθούμε αυτών των ε, αρμοδιοτήτων και να τι αναθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή. Επίση, θεωρούμε ότι θα έχει ψηλό κόστο διοικητικό η αρχή αυτή, θα επιβαρύνει τα κράτη-μέλη. Το πεδίο αρμοδιοτήτων της σχεδιαζόμενης νέας αρχής είναι ασαφές. Υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της μετά από σχετική αξιολόγηση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η νέα αρχή θα επιδιώξει να αναλάβει περαιτέρω αρμοδιότητα. Αυτό συμβαίνει με κάθε νέα αρχή, με κάθε νέο οργανισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε για πολιτικές που δεν χρειάζεται να αρμονιστούν περαιτέρω, όπως ε, το πώς καθορίζονται τα μισθολόγια. Για να ολοκληρώσω, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακόμη μια απόπειρα να ε, αντιμετωπίσει θέματα γραφειοκρατίας που οι ίδιες τις οδηγίες έχουν προκαλέσει. Δηλαδή, αντί να ε, απαλείψει την γραφειοκρατία που έχει δημιουργήσει η ίδια επιτροπή μόνη τη με άλλο τρόπο, ψάχνει να δημιουργήσει μια νέα αρχή. Το μόνο που μου αρέσει ε, από την ε, όλη ιδέα είναι η συντομογραφία ΕΛΑ, το όνομα. και μια ερώτηση τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ωφέλει Σκοπεύεται να ε, προκύψουν πιστεύω ότι θα προκύψουν από αυτή την αρχή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες προσπάθειες για την συμπλήρωση εντύπων, περισσότερη γραφειοκρατία ενδεχομένως. Ποιο είναι το κόστος για τα κράτη-μέλη και ποιο από το κόστος αυτό θα καλύπτεται σε προηγούμενη φάση. θα έχει μόνο συντονιστικό ρόλο η αρχή αυτή ή θα αναλάβει και αρμοδιότητες των εθνικών ελεγκτών. Και έχω και ερώτηση για την έδρα της αρχής. Ευχαριστώ κύριε Σλοτόφσκι. Ε, επειδή είμαι και εγώ σκιώδης εισηγήτρια, κύριε Λιεζουά, σας ευχαριστώ για την εισηγήσή σας είναι ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερη προσοχή. Εάν η αρχή αυτή ιδρυθεί όντω, πρέπει να κοιτάξουμε να είναι αποτελεσματική. Αποτελεσματική, διότι ιδίω στον τομέα των οδικών μεταφορών, να θυμίσω ότι στου αυτοκινητοδρόμου τη Ευρώπη έχουμε καθημερινά 2 εκατομμύρια. 2 ε, εκατομμύρια τουλάχιστον ε, που ε, οδηγούς φορτηγών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η αρχή να λειτουργεί και να έχει και πραγματικό αντίκτυπο. Η πρώτη ερώτηση που με απασχολεί είναι τι θα γίνει αν μια κυβέρνηση δεν θέλει να συνεργαστεί. Τι θα την κάνουμε. Τι θα την κάνουμε την εθνική της αρχή. Τι θα γίνει στην πράξη. Θα επιβληθούν κυρώσεις. Προς στιγμήν δεν έχουμε ιδέα. Δεύτερη ερώτηση που μου φαίνεται εξίσου σημαντική. Πρόκειται για μία συνένωση στην αρχή αυτή των προηγούμενων αρχών και οργανισμών που γνωρίζαμε. Ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Επαγγελματικής Υγείας, ώσα. Ε, ε, θα Έχουμε την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το Ίδρυμα για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας. αυτά τα τρία, οι τρεις οργανισμοί, οι τρεις ενώσεις και ιδρύματα θα ενοποιηθούν στην νέα αρχή ή πώς θα διαρθρωθεί η πως θα διαρθρωθει η εργασια τους. Επίσης, η αρχή αυτή φαίνεται να ασχολείται περισσότερο με τα θέματα απασχόλησης και εργασίας. Εγώ διαρωτώ με, στην πράξη, τι θα γίνει στα κράτη όπου οι αρχές που ασχολούνται με την απασχόληση ή οι επιθεωρητές εργασίας είναι θύματα ε, των δημοσιονομικών περικοπών ε, ε, τα τελευταία χρόνια σε υψηλά επίπεδα κιόλας πώς θα ε, διαρθωθεί αυτή η συνεργασία με τους περιορισμένους πόρους των κρατών Και ε, έπειτα για μένα αυτή η αρχή δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια πλατφόρμα ανταλλαγή καλών πρακτικών. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον τότε, δεν είναι μια ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ εθνικών εμπειρογνωμόνων ο σκοπό. Νομίζω ότι η ευρύτερη θεώρηση τη αρχή αυτή θα είναι να πρέπει να φροντίσει την, ε, για την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό είναι η ουσία. Να επιβάλλει κυρώσει να επιβλέπει την σωστή εφαρμογή του δικαίου. Και τέλος να πω και κάτι ακόμη λέτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρέπει στην αρχή αυτή ένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων για την εργασία, των ε, περιορισμών που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις κτλ. Αλλά επί τη ουσία, η ερώτησή μου εμένα είναι ποιο θα προστατεύει του καταγγέλλοντε, αυτού που ε, θα καταγγέλουν ένα πραγματικό πρόβλημα σε μια επιχείρηση. Η αρχή αυτή, τι ακριβώ θα κάνετε. Και δεύτερο στοιχείο, και αυτό θέλω να το πω, διότι αυτό θα κάνει την αρχή να έχει κάποια χειροπιαστή αρμοδιότητα και κάποια βαρύτητα. Διότι επαφιέται στη κρατική ευκαιρία των κρατών μελών. Όμω, για να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αρχή πρέπει να έχει και κάποιο ρόλο ελέγχου. Εάν δεν τον έχει, ε, Ποιο λοιπόν θα την αναλάβει αυτή την ευθύνη του ελέγχου, εφόσον τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει τίποτε ω τώρα και δεν βλέπω γιατί να αλλάξουν τη στάση του. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει νόημα να δημιουργηθεί άλλη μια αρχή απλώ για να υπάρξει και να χαρούν κάποιοι. Αυτό είναι και το γενικότερο δράμα των αρχών και των οργανισμών. Να σα βοηθήσουμε, κύριε Λιεζόα, βέβαια, αλλά για να σα βοηθήσουμε πρέπει η αρχή, ο οργανισμό να έχει ρόλο αυτό συγκεκριμένο και να είναι αποτελεσματική. Δηλαδή με την τεχνολογική και ψηφιακή ε, επανάσταση θα αλλάξουν όλες αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες και οι έλεγχοι. Οι εξελίξεις θα μας προλάβουν. Ε, πρέπει να ε, ξεκινήσει τώρα η προσπάθεια για την αρχή αυτή ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μπιλμπάο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έγινε κάποιο λάθος σχέση με το πότε ζήτησα τον λόγο. Πρόκειται λοιπόν για μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να είναι απαραίτητη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και αρκετές ε, αμφιβολίες σχετικά με τις αρμοδιότητες τις οποίες θα θέλαμε να έχει η υπηρεσία αυτή και τις οποίες δεν βλέπουμε να παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσα να σας τις περιγράψω το θέμα των μεταφορών σαν παράδειγμα. Προβλέπεται ε, στα πλαίσια της οδηγίας για τις αποσπάσεις ένας μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να ζητήσει από τα άλλα κράτη-μέλη ε, πληροφορίες, ε, υπάρχει ένα σύστημα δηλαδή καθορισμένο ε, για την ενημέρωση. Ένας μηχανισμός λοιπόν διακρατικός ad hoc δεν ξέρω πώς θα καλύψει τις αρμοδιότητες ή θα ενταχθεί στις αρμοδιότητες του νέου συστήματος. Αναφερθήκατε επίσης και στον κοινωνικό πυλώνα. Ο κοινωνικός πυλώνας είναι κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί στο Γκότεμπορκ το 2017 και υπήρξε μία σειρά συστάσεων προορισμένων προς τα κράτη-μέλη. Όταν εντάξουμε σε αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα αυτές τις συστάσεις, ποιες είναι οι αρμοδιότητες τις οποίες θα έχει η προτινόμενη υπηρεσία στον κοινωνικό πυλώνα. Προβλέπεται επίσης ένα διπλό σύστημα στο πακέτο για την κινητικότητα, περιλαμβάνεται σε πολλές εκθέσεις και παρουσιάσεις. Και σε σχέση τώρα και κυρίως με τους στόχους, η πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αυτό είναι κάτι αρκετά εύκολο. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης οι πληροφορίες για την εργασία από κάθε κράτος μέλος και κάθε τομέα ε, για την συνεργασία. Ποιος θα συνεργαστεί όμως. Εγώ είμαι υπέρ επαναλαμβάνω λέει η κυρία Μπιλμπάου. Και υπερασπιστήκαμε στο πακέτο έτσι και αλλιώ για τις μεταφορές, τις μονοπευθυντικές θηρίδες, όπως επίσης και τη σωστή αμοιβαία ενημέρωση. Νομίζω ότι και εκεί είναι ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία υπηρεσία τώρα. Είναι σαφές επίσης ότι δεν θα πρέπει να αναλάβουν τις αρμοδιότητες ε, και τις εξουσίες ε, των εθνικών αρχών. Πώς όμως θα συνεργαστεί με αυτές τις, εθνικές αρχές και τι δυνατότητα έχουν ε, να ζητούν αυτές τις, αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι δεν είναι, απλό, δεν είναι μόνο το να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα συλλέγει πληροφορίες. Θα πρέπει να πάει ακόμα περισσότερο, να απαιτεί την εφαρμογή, να... Ταυτόχρονα δεν θα έχει καμία δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και δεν θα έχουν και τα κράτη-μέλη καμία υποχρέωση να ενημερώνουν και να δίδουν απαντήσεις στην υπηρεσία αυτή, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα με περισσότερες αρμοδιότητες στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής. Λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε ένα περαιτέρω βήμα. Και δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι και εμείς σε επίπεδο κοινοβουλευτικό να σας βοηθήσουμε να κάνετε κάτι το πιο σταθερό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπιλμπάου. Κυρία Βονταλόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι καρπός ε, μακρών αγώνων του Κοινοβουλίου για την καλύτερη εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και την παράσπιση των εργαζομένων στο σύνολό τους. Ε, και χάρη στην αφοσίωση των βουλευτών και την προσπάθεια για πρόθεση στην κοινωνική Ευρώπη έγινε αυτή η πρόταση. Λέω δεν θα έχει δει ποτέ το φως της ημέρας και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Η πρόταση είναι για τέλη 18 να τεθεί σε ισχύ και το 2019 να αναλάβει καθήκοντα αυτή η νέα αρχή. Δεν ξέρω αν αυτό σα φαίνεται ρεαλιστικό. Έχοντα υπόψη η νομοθετική συμφόρηση, επειδή βρισκόμαστε στο τέλο τη θητεία, στο μέσο των μεταφορών, να εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και στο πεδίο εφαρμογή, αλλά είναι αρκετά θολά τα όσα λέγονται για τι αρμοδιότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία στον τομέα αυτό και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Μπιλμπάου επ' αυτού. Πώς θα γίνει η διασύνδεση μεταξύ αυτής της αρχής και της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Μητρώου Δικών Μεταφορών. Στην πρόταση ε, επίσης λέγεται ότι δεν θα έχει ε, κάποια προνόμια η, Επιτροπή, ε, η Αρχή Εργασίας για να μπορεί να ασκεί πίεση στις εθνικές αρχές. Αυτό είναι περιορισμός. Αν δεν μπορεί επίσης πάλι κάποιες αρχές, σε κάποιες εθνικές αρχές αν υπάρχει σύγκρουση ή υπάρχει ζήτημα ανταλλαγές πληροφοριών. Όλα αυτά τα συζητάμε και στο πακέτο για την κινητικότητα. Δεν είναι κακό ε, που έγινε αυτή η πρόταση, πρέπει όμως να γίνει πιο ε, στεναρή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαχ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω τη σημασία της ε, πρότασης. Το είπαν όλοι οι συναδελφοί μου ανεξαιρέτως ε, και <clears throat> το υπογράμμισαν στις μεταφορές ιδίω νομίζω ότι θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Θα είχε προσταμένη αξία δημιουργία αυτής της αρχής. Ποια είναι ο κίνδυνος που βλέπω να επιφορτιστεί με πάρα πολλά καθήκοντα η Ευρωπαϊκή αυτή αρχή. Ε, το είπε νομίζω και κάποιοι προλαλήσαντες ε, ότι δηλαδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την εφαρμογή της νομοθεσία και θα είναι ουσιαστικά ένας ξεδοντιασμένος τίγρης ε, η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όμως ε, πρέπει να έχει ε, την απαραίτητη δύναμη. Πιστεύω λοιπόν ότι η Καρίμα ε, μας έδωσε τη σωστή ε, κατεύθυνση. Έχω σε ένα ερώτημα. Η συνεργασία μας ε, με την αρχή που ήδη υπάρχει, πώς θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε στην πράξη, τι γίνεται και με τις αρχές των κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα ο εισηγητής κάπως με απογοήτευσε. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι δεν θα πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι εθνικές αρμοδιότητες. Αυτό όμως για μένα είναι κλειδί. Η αρχή εργασίας θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες για να μπορεί να επιβάλλει κάποια πράγματα στα κράτη-μέλη. Αλλιώς ε, δεν έχουμε ε, τη δυνατότητα να ε, επηρεάσουμε τις επιχειρήσεις. Είμαι υπεύθυνο ε, για το πακέτο, για το, σιδερο, τέταρτο πακέτο και την Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Σιδηροδρόμων. Ε, επί καιρό αγωνιστήκαμε. Αν δεν θέλουν να υπάρχει μια πραγματική αρμοδιότητα η οργάνωση εργασίας αυτή, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα, το θέμα της επιβολής, της εφαρμογή, είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρικέ έχει τώρα το λόγο. Δεν θέλω να επισέλθω στη συζήτηση για τον οργανισμό, αλλά έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο βαθμό που δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Αρμοδιότητα στις συνθήκες για το θέμα. Υπάρχει έστω και κάποια ελάχιστη δυνατότητα με προτάσει του Κοινοβουλίου να μπορεί να έχει κάποιες εκτελεστικές αρμοδιότητες αρχή αυτή άκουσα την πρόταση Κομισιόν και νομίζω ότι ευθυγραμμίστηκε με τις συνθήκες. Είναι δηλαδή σόφρον. Ένα έργο συντονισμού, τεκμηρίου, ανταλλαγών κτλ. κτλ. Δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση αυτή η αρχή ε, να διαιτητεύσει ή να επιβάλλει ή να επιβάλλει ε, κυρώσεις ε. Εμείς θα θέλαμε πιο αποτελεσματικά μέτρα, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Ρικέ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο. Ε, υπάρχουν όμως πάρα πολλές ερωτήσεις. Να απαντήσετε εσείς κύριε Λίζου. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Βέβαια θετικές είναι οι παρατηρήσεις ε, ως επιτοπλίστων και νομίζω ότι θα ενισχύσουν ουσιαστικά οι προτάσεις αυτές ε, τις εξουσίες και αρμοδιότητες της αρχής εργασίας. Ε, προσπάθησα να σχολιάσω στα αγγλικά τώρα ο κύριος Λεζουά για αυτές τις ε, δράσεις ή λειτουργίες. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που θα είναι αρμοδιότητα της αρχής αυτής. Είναι αντικείμενο ε, ε, το οποίο συζητά και η Επιτροπή Απασχόληση, Εργασία ή Απόσπαση Εργαζομένων. Όλε αυτέ τι δραστηριότητε ε, τώρα θα είναι αρμοδιότητα τη αρχή εργασία. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση γιατί έχουμε ε, πλέον μία αρχή αρμόδια Σε ό,τι αφορά πιθανέ αλληλεπικαλύψει με τι εθνικέ αρχέ, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη και οι εθνικέ ε, αρχέ επιβολή νομοθεσία διατηρούν τι βασικέ του αρμοδιότητε, που είναι η επιβολή τη νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία θα συμπληρώνει τη δράση των εθνικών αρχών. Δεύτερο, έδρα. Είμαστε στις ε, αρχές της συζήτησης ε, σε επίπεδο Συμβουλίου. Υπάρχει μια κοινή προσέγγιση του 2012 μεταξύ των κοινών των τριών θεσμικών οργάνων αποφασίστηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί από τα κράτη-μέλη. Ήταν κάπως επιφυλακτικά στα σχολεία του κ. Λοτόφσκη και το σημειώνω αυτό. Δεν θα υπάρχει ανάγκη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών γιατί ήδη, εργάζεται, ε, ήδη μάλλον ε, η συνεργασία λειτουργεί πολύ καλά. Δεν αληθεύει αυτό. Υπάρχει για την υποχρέωση των κρατών μελών να οργανώ έξι συντονισμένου ελέγχου. Γι' αυτό απαιτείται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Μόνο τα μισά κράτη-μέλη συνεργάζονται και μπορούν να οργανώσουν του ελέγχου αυτού. Άρα δεν ισχύει ότι υπάρχει ήδη πολύ καλή συνεργασία. Τώρα, αν θα υπάρξει προσθέμενη αξία για τι επιχειρήσει και δίτε ΜΜΕ, φυσικά και θα υπάρχει, γιατί αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε είναι φυγή εφαρμογή ουσιαστικά τη νομοθεσία, ώστε από τη μία να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ε, το βάρο ε, των επιχειρήσεων, απλουστεύοντα τι διατυπώσει και το διοικητικό ε, και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια πιο ευφυή ε, εφαρμογή της νομοθεσίας βελτιώντας τη συνεργασία ακριβώς μεταξύ των κρατών μελών. Κυρία Πρόεδρε, στα γαλλικά τώρα. Ε, με βομβαρδίσατε με ερωτήσει εσεί, κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο λέτε τι θα γίνει αν τα κράτη-μέλη θέλουν να συνεργαστούν. Το είπα και στην παρουσίασή μου, πράγματι δεν υπάρχει πραγματική αρμοδιότητα η, Επιτροπή, η αρχή αυτή να επιβάλλει κάτι règlement si des États membres, euh, par Αν δεν ε, θέλει κάποια να συμμετέχει στους κοινούς ελέγχους, θα πρέπει να ε, προβάλλει ε, βάσιμους λόγους για κάτι τέτοιο. Ε, δεν υπάρχει πράγματι, πραγματική αρμοδιότητα και εξουσία για επιβολή κάποιων όρων. Τώρα, αν υπάρχει κάποια επίπτωση για άλλους οργανισμούς. Σαφώς και όχι. Θα πρέπει όμως να συνεργαστεί με αρκετού άλλους οργανισμούς αυτή η νέα αρχή. Και το είπα και στην παρουσίασή μου, ήδη υπάρχει ένα advisory group το οποίο θα προετοιμάσει τη σύσταση και συγκρότηση αυτή τη ε, αρχής και εκεί θα υπάρχουν διάφοροι stakeholders οι οποίοι θα συμμετέχουν. Ήδη ιδέα μεταξύ αυτών είναι οι φυστάμενοι οργανισμοί για να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή αυτή αρχή εφόσον συσταθεί και όταν συσταθεί μιλήσετε για το πρόβλημα έλλειψη πόρων στα κρατημέλη. Αυτό αληθεύει και το έχουμε ε, συμπεριλάβει στις αναλύσεις μας για το πρώτο πακέτο κινητικότητας. Όμως πρώτα απ' όλα είναι ευθύνη των κρατών μελών. Τουλάχιστον η αρχή αυτή εργασία θα μπορούσε να επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων ακόμη και αν αυτοί μειούνται στα κρατη ε, σωστά είπατε ότι δεν θα πρέπει να είναι άκαμπτη, αλλά να εξελίσσεται μια τέτοια αρχή εργασίας. Και ναι, συμφωνώ. Και προβλέπεται αναθεώρηση πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού. Βέβαια, εξέλιξη δεν θα πει ότι θα πρέπει να υπάρχει ασάφεια στην αρχή, και αν διαβάσετε το σχέδιο κανονισμού και την ετολική σκέψη 8, στη γάμα δελτα μούβ εμείς αυτό που θελήσαμε είναι ήδη ε, να υπάρχει σαφής ένδειξη ε, για τις ε, δραστηριότητες και τους τομείς δράσης. Έχουμε το 1071 κανονισμό για την πρόσβαση ε, στη, στα διάφορα επαγγείλματα, πολέμηση, δηλαδή των γραμματοκιβωτίων, ε, το ιδίων γραμματοκιβωτίων. Επίσης ε, υπάρχει το πακέτο κινητικότητας 1 που περιλαμβάνει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Και υπάρχει δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να να επιτρέψει μεγαλύτερη συνεργασία. Υπάρχουν δύο σκύλες. Ένα άλλο ερώτημα. Ποιε θα είναι εξουσίε της ε, αρχή εργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμοδιότητε τη Ένωση δεν είναι ισχυρέ. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να μια διάκριση. Πράγματι υπάρχει κοινωνικό τομέα που είναι αρμοδιότητα των συναδέλφων από την ΔΕΛΤΑ Απασχόληση και εκεί πράγματι η αρμοδιότητα είναι μεικτή μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εδώ είμαστε στον τομέα της εργασίας. Όμως, αν ε, δούμε τι γίνεται στον τομέα των μεταφορών, κυρίως των οδικών μεταφορών, έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Εγώ θα ότι έχουμε και αποκλειστική μάλιστα αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ισχυρή λοιπόν αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή λοιπόν θα έχει και αυτή αρμοδιότητες. Αυτά και κυρίως από την κυρία Μπιλμπάου. Σημειώνω τις επιθυμίες σας και η κυρία Επίσης είπε κάποια πράγματα που τα λαμβάνω υπόψη. Θέλετε, είπατε, να είναι πιο ισχυρή η αρχή εργασία, να μπορεί να επιβάλλει, να εξαναγκάζει τι εθνικές αρχές να προβούν σε κάποια μέτρα. Και η θεσμική συζήτηση που θα ακολουθήσει μεταξύ κοινόβουλου και συμβουλού θα μας δείξει που θα βρεθεί η χρυσή τομή τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λίζουα. Στη φάση αυτή βρισκόμαστε ακόμα στο επίπεδο των συζητήσεων και θα πρέπει να, να προβλέψουμε ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων για αυτή την αρχή που να μην ε, συμπίπτει με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οπότε πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μα διαθέσατε το χρόνο σα. Και τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Διάλειμμα γιατί είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από ό,τι προβλεπόταν. Όχι πολύ. Όχι πολύ. 20 λεπτά, έτσι. Για να γνωρίζετε. Μετά Ακούστε με παρακαλώ προσεκτικά. Στις 11 όλα θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπό Μπούλτς για όλα τα θέματα που αφορούν την κινητικότητα, τις μεταφορές, ε, τα πάντα, στις 11 εδώ και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κάμερες. Και βεβαίως προσκεκλημένοι είστε όλοι οι βουλευτές. Σε 20 λεπτά λοιπόν θα τα πούμε. Σε hors caméra.